Θα μπορούσαμε παρακαλώ να ανοίξουμε τις πόρτες, να κάνουμε πάλι δημόσια τη συνεδρίαση. We are in a hurry. Βιαζόμαστε. Mm-hmm. Ah, wir kommen. oh, yeah, σας ευχαριστώ. Σας ε, ζητώ συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση. Και θα περάσουμε στο σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης, συστημικά προβλήματα στην επιμερισμένη διαχείριση των διαθερωτικών ταμείων στη Ρουμανία και την Ουγγαρία. Καλέσαμε την ε, τον εκπρόσωπο της ε, Επίτροπου Κρέτσου, κύριο Λεμέτ. Υπάρχουν προβλήματα και στις δύο αυτές χώρες σχετικά με την ε, διαχείριση των ε, ταμείων. Έχουν ε, μεγάλα προβλήματα. Και η φυστάμενη νομοθεσία σε ό,τι αφορά τα θέματα διαφθοράς πολιτικών ή διοικητικών ε, θα αλλάξει. Ε, γνωρίζετε εσείς καλύτερα την κατάσταση στη Ρουμανία. Έχουμε και έναν εκπρόσωπο της Ουγγαρίας εδώ. Θα θέλαμε λοιπόν να μας κάνετε μία εκτίμηση της κατάστασης. Πώς επηρεάζονται τα ε, ταμεία και η χρήση τους εξαιτίας αυτών των δυσκολιών και πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση στη Βουδαπέστη για την Ουγγαρία, αλλά και στη Ρουμανία υπάρχουν συστημικά προβλήματα. Ενδεχομένως και στην Ουγγαρία να υπάρχουν συστημικά προβλήματα. Είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν πολλά χρόνια. Από το 2011 μάλιστα έχουμε επίγνωση της κατάστασης όπου επισκεφτήκαμε τέτοιες περιπτώσεις, επισκεφτήκαμε κάποια έργα και είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια. Αλλά θα δώσω σε εσάς το λόγο για, όποια, για τη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Θα κάνω ό,τι μπορώ προκειμένου να απαντήσω τα δύο συγκεκριμένα θέματα τα οποία μόλις ε, υπενθυμίσατε και περιγράψατε και πάλι. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τη Ρουμανία και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια αλλαγή στην νομοθεσία. Είναι πολύ βολική η στιγμή, διότι αυτή την εβδομάδα, μάλλον την προηγούμενη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον πιο προσ... την πιο πρόσφατη έκθεση συνεργασίας και μηχανισμού επαλήθευσης για τη Ρουμανία αφενός και για τη Βουλγαρία αφετέρου. Εγώ δεν είμαι υπεύθυνο ε, για την έκθεση αυτή. Ο πρώτος αντιπρόεδρος Τίμερμανς ε, είναι αρμόδιος. Επομένως, ε, για το θέμα αυτό θα αναφερθώ κυρίως στα όσα έχει πει σαφέστατα κατά την παρουσίαση της πιο πρόσφατης έκθεσης και ε, του τι περιλαμβάνει ε, η έκθεση για τη Ρουμανία όσον αφορά αυτά τα οποία διαπιστώσαμε για τη Ρουμανία τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Η γενικότερη αξιολόγηση που γίνεται στην έκθεση για τη Ρουμανία είναι ότι υπάρχει συνεχής συνολική πρόοδος. Ταυτοχρόνως βεβαίως δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε και το γεγονός ότι το βασικό μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι επιμένουμε ότι αυτή η πρόοδος ε, πρέπει να γίνει ανεπιστρεπτή. Και αυτή είναι ορολογία η οποία χρησιμοποιείται ε, συγκεκριμένα για τη Ρουμανία. Για τα δύο ε, σχέδια κατεπίγουσας διαταγής που αναφέραμε, Υπάρχουν δύο εδάφια στην ενέκθεση του Μηχανισμού Συνεργασίας ε, και Επαλήθευσης που ε, αναφέρονται στο θέμα αυτό. Το πρώτο λέει ότι τα δύο κατεπήγοντα κείμενα τα οποία δόθηκαν για διαβούλευση από την ε, ε, ε, κυβέρνηση θα οδηγήσουν σε αντίθεση για την ε, διαφθορά και την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Και η δεύτερη αναφορά σε αυτές τις εξελίξεις για αυτά τα διατάγματα είναι στη σελίδα 13 που λένε ε, σαφέστατα ότι οποιοδήποτε τελικό κείμενο των δύο διαταγμάτων που έχουν τεθεί κατεπηγόντως ε, προς ε, συζήτηση θα πρέπει να εξεταστούν υπ' αυτό το πνεύμα. Και το υπ' αυτό το πνεύμα αναφέρεται σε μια πιθανή ανάγκη επαναξιολόγησης της προόδου που έχει ε, επιτελέσει η Ρουμανία. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγω εγώ από αυτό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί το θέμα στενά ε, το γεγονός ότι το θέμα αυτό εμπίπτει πλήρως εντό της εντολής ε, της συνεργασίας και επαλήθευσης και του σχετικού μηχανισμού και οποιαδήποτε νέα νομοθεσία τεθεί σε εφαρμογή στη Ρουμανία, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή, θα αξιολογηθεί βάση του μηχανισμού διόρθωσης και επαλήθευσης. Με ρωτήσατε κατά πόσον διαβλέπω κάποια άμεση ε, σχέση με τη διαχείριση των, των κονδυλίων. Πρώτον, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσουμε τις νομικές εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια νομική εξέλιξη, αλλά ε, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ των όσων εμπίπτουν στη διαδικασία του μηχανισμού συνεργασίας και επαλήθευσης και μεταξύ των όσων έχουν συσταθεί για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς εντός των κανόνων των διαρθρωτικών ε, ταμείων. Όπως ξέρετε, έχουμε αναβαθμίσει σημαντικά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου για την παρούσα δημοσιονομική περίοδο και για τη Ρουμανία ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια ανάθεση ε, συστημάτων μηχανισμού και ελέγχου και αυτό σημαίνει ότι δεν έχει γίνει κάποια υποβολή για πληρωμή. Υποστηρίζουμε τη Ρουμανία όσο μπορούμε και θα την υποστηρίξουμε και μέσω ε, ατομικών επιχειρησιακών προγραμμάτων. υπάρχει μια συγκεκριμένη σειρά όρων που θα πρέπει να εφαρμοστούν εκ των προτέρων για τους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, τις δημόσιες προμήθειες που είναι πάρα πολύ απαιτητικοί για τη Ρουμανία. Η Ρουμανία ακόμα τα επεξεργάζεται, δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος ε, όσον αφορά τη δημιουργία ικανοτήτων ε, και μέσω της δημιουργίας ε, μια εθνική υπηρεσία για τις δημόσιες προμήθειες. Θα ξεκινήσουν δύο πολύ συγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα για χρηματοοικονομική υποστήριξη και ε, θα υποστηρίξουν τη Ρουμανία σε όλο αυτό το διάστημα προκειμένου να μπορέσει να αναβαθμίσει περαιτέρω και ε, τις δικαστικές της δυνατότητες και τις δυνατότητές της ε, σε θέματα δημοσίων προμηθειών. Σε γενικέ γραμμέ λοιπόν για τη Ρουμανία θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε ένα πολύ συνεργάσιμο εταίρο, αλλά λόγω του πολύ υψηλού επίπεδου απαιτήσεων που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να ξεκινήσει η παρούσα περίοδος, ακόμα ε, εκκρεμούν πάρα πολλά πράγματα προκειμένου να μπορέσει τελικά να ε, καθορίσει η Ρουμανία τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου και να είμαστε και εμείς ικανοποιημένοι ότι η Ρουμανία ε, διαθέτει πλέον ένα εύρωστο σύστημα δημοσίων προμηθειών ε, για την παρούσα περίοδο. Να περάσω τώρα στην Ουγγαρία. Εκεί αναφερόμαστε στα πιο πρόσφατα γεγονότα Λάβαμε μια έκθεση από την Όλαφ στις 6 Δεκεμβρίου του 2016. Πολύ σωστά αναφερθήκατε στο χρόνο που χρειάστηκε προκειμένου η Όλαφ να εκπονεί την έκθεση. Ε, Αφορμή για την ε, έναρξη της έκθεσης της Όλαφ ε, ε, δόθηκε το 2012 όταν και το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο προώθησαν πληροφορίες στην Όλαφ για την γραμμή μετρό 4 της Βουδαπέστης και Η Όλαφ ε, έκανε μια μακρά έρευνα η οποία από ό,τι γνωρίζουμε σχετίζεται και με την ανάγκη ε, να μπορέσει η Όλαφ ε, να έρθει σε επαφή με αρκετές δημόσιες αρχές σε διάφορα κράτη-μέλη. Δεν ήταν αποκλειστικά στην Ουγγαρία και σχετίζεται επίσης και με το γεγονός ότι η Όλαφ εξέτασε συνολικά πάνω από 100 συμβάσεις. Μετά από την έκθεση λοιπόν που λάβαμε, Ακολουθήσαμε αμέσως τη συνήθεια διαδικασία για το θέμα αυτό, δηλαδή εξετάσαμε την έκθεση γιατί σε, στην Επιτροπή Αναστολών Διακοπών και Οικονομικών Διορθώσεων που αποφάσισε να παραπέμψει αυτή την έκθεση στις Ουγγρικές Αρχές για να τους δώσει τη δυνατότητα να ε, κάνουν παρατηρήσεις. Η έκθεση ε, εστάλει λοιπόν πριν από το τέλος του προηγούμενου έτους στις Ουγγρικές Αρχές, οι οποίες εντωμεταξύ ζήτησαν και έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν, να δοθεί η έκθεση στην ουγγρική γλώσσα και μαζί με την Όλαφ ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μπορέσει να δοθεί μετάφραση στην Ουγγαρία το συντομότερο δυνατόν. Όπως αντιλαμβάνεστε βεβαίως, ε, πρόκειται για ογκώδη έκθεση πολύ τεχνικής φύσεως, επομένως η μετάφραση θα καθυστερήσει λίγο, αλλά ε, πιστεύουμε ότι το αργότερο το Μάρτιο θα μπορέσουμε να του στείλουμε αυτή την έκθεση uh, uh, uh, για να έχουν και χρόνο να μας στείλουν από εκεί και πέρα να παρατηρήσεις και να μπορέσουμε να δούμε ε, τις παρατηρήσεις τους και να καταλήξουμε σε μια ορεστική θέση επί της υποθέσεως αυτής και την ανάγκη να ε, υπάρξουν ίσως ε, οικονομικές διορθώσεις και επιστροφές ποσών. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω ήδη από σήμερα είναι ότι το πρόγραμμα αυτό στο οποίο ανήκει το έργο του Μετρό της Βουδαπέστης ε, για τη γραμμή 4 δεν θα κλείσει και δεν θα λάβουμε οριστική η τελεσίδικη απόφαση όσον αφορά τις οικονομικές διορθώσεις και σε κάθε περίπτωση θα βασιστούμε μόνον στα γεγονότα για να καταλήξουμε σε κάποια τελική απόφαση και δεν θα μας επηρεάσει το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν συνέπειες επειδή βρισκόμαστε στο τέλος ε, μιας οικονομικής περίοδου που σημαίνει ότι ε, μπορεί οι διορθώσεις αυτές ε, να μην μπορούν να αποζημιωθούν από άλλες δαπάνες. Θα ακολουθήσουμε μια πάρα πολύ αυστηρή και συνεκτική γραμμή για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε κυρίως στην ολοκλήρωση των προγραμμάτων να έχουμε μηδενική ανοσυχή για τη διαφθορά και την απάτη. Ευχαριστώ πολύ. Σα Σας ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Γνωρίζουμε πώς δεν είναι εύκολα τα πράγματα, ειδικότερα στη Ρουμανία, αλλά εσείς ε, τι νομίζετε, θα μπορούσαμε να στείλουμε ε, μέσω αυτών των ενεργειών και ένα μήνυμα στις υπόλοιπες χώρες, να μάθουμε από τα προβλήματα. Ε, τώρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση της καταστάσεως ε, στη Ρουμανία. Θα ήθελα να αναφέρω δύο-τρία στοιχεία και να αναφερθώ σε κάποιες πτυχές που εξετέθησαν για να είναι όλα ξεκάθαρα για όλους. Η έκθεση του Μηχανισμού Συνεργασίας είναι άκρος θετική όσον αφορά τη Ρουμανία και δείχνει την πρόοδο που επετέλεσε η Ρουμανία στα πλαίσια του μηχανισμού συνεργασία και επαλήθευση και δείχνει ότι έγιναν πολλέ πρόοδοι και πρόοδοι που δεν μπορούν να αντιστραφούν. Υπάρχουν φόβοι βέβαια, όχι μόνο στι Βρυξέλλες αλλά και στη Ρουμανία, πραγματικοί φόβοι που σχετίζονται με προγράμματα ε, κατάσταση ανάγκης κατεπήγοντα προγράμματα που συζητούνται δημοσία. Τα, τα διατάγματα που αφορούν το συνταγματικό δικαστήριο της Ρουμανίας που αφορά τον ποινικό κώδικα, διότι κάποια άθρα του ποινικού κώδικα δηλώθηκαν ότι είναι αντισυνταγματικά από το συνταγματικό δικαστήριο της χώρας. Λοιπόν, τα κατεπήγοντα διατάγματα ακολουθούν την απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου, δηλαδή ενσωματώνουν στην ομοθεσία, αυτές τις διατάξεις ή κάνουν την, ε, την ομοθεσία να εναρμονίζεται με την απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου. Είναι τεχνικής φύσεως υποχρεώση της ε, ρουμανικής κυβερνήσεως. Από την άλλη πλευρά έχουμε την κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές της Ρουμανίας ε, είναι πολύ κακές οι συνθήκες ε, κράτησης λόγω υπερπληθισμού και πολλές αποφάσεις των ε, του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουν ληφθεί υπέρ των κρατουμένων και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ασκεί πιέσεις ούτως ώστε ο αριθμός των κρατουμένων να μειωθεί αναφυλακή είτε μέσω οικοδόμησης νέων φυλακών ή μέσω άλλης λύσεως. Θα πρέπει οι συνθήκες κρατήσεως να ε, πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Οι φόβοι συνδέονται με το ότι τα διατάγματα αυτά που υπογράφονται θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και υπέρ εκείνων που είναι κρατούμενοι λόγω διαφθορών. Το ποσοστό λοιπόν όμως εκείνων που κατηγορούνται για πράξεις που καλύπτονται τα διατάγματα και που είτε εκδικάζεται η απόφασή τους είτε βρίσκονται στη φυλακή είναι το 1,6% των υποθέσεων. Αλλά παραμένουν φόβοι και η καταπολέμηση της διαφθοράς θα πρέπει να είναι ο βασικός μας ε, στόχος. Όχι μόνο όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς πόρους αλλά εν γέννη όταν πρόκειται για τις επενδύσεις στη Ρουμανία, για το δημόσιο χρήμα εν γέννη. Βελτιώθηκε η κατάσταση όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι έχουμε καλό σύστημα εκεί. Η κυβέρνηση της Ρουμανίας είναι διαθέσιμη να προωθήσει την εύρυθμη λειτουργία των πραγμάτων. Κατά το παρελθόν πολλές συμβάσεις ανετίθεντο χωρίς να ακολουθούνται οι σωστές και αναγκαίες διαδικασίες. Το ότι αυτά τα δύο διατάγματα συζητούνται δημοσίως και χτες μάλιστα Δευτέρα οργανώθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνη δημόσια συζήτηση και το ότι τα δύο προγράμματα και τα δύο διατάγματα συζητηθούν στο Κοινοβούλιο είναι θετικό. Και όσον αφορά το διάταγμα για τη συλλογική χάρη, αυτός ο όρος χάρη κάνει κάποιον να σκέφτεται πολιτικούς που κατηγορούνται για διαφθορά. Δεν πρόκειται για αυτούς, αλλά δεν πρέπει να λησμονήσουμε ότι υπάρχει μεγάλη ευαισθησία στη Ρουμανία, στη ρουμανική κοινωνία ο κόσμος διαδήλωσε την Κυριακή και πρέπει να πούμε ξεκάθαρα στους εξωτερικούς εταίρους μας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους και στους Ρουμάνους ότι εδώ δεν μιλάμε για τους ε, πολιτικά υπεύθυνους, τους διεφθαρμένους πολιτικούς. Πρόκειται για δύο άλλα θέματα. Πρόκειται για το Συνταγματικό Δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ασκούν πιέσεις επί της κυβερνήσεως για να ξεκαθαριστεί η κατάσταση. Στη Ρουμανία η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί πάντα προτεραιότητα και καμία κυβέρνηση ανεξάρτητα από το πολιτικό της χρώμα δεν θα κάνει λιγότερες προσπάθειες. Και έχω και μία ερώτηση που απευθύνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, οι ευρωπαϊκοί πόροι πώς μπορεί να διατεθούν, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν, πότε η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα θα σταματήσει. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιο προσανατολισμό χρονικό, διότι πέρασαν ε, χρόνια τώρα από όταν ξεκίνησε η περίοδος και το επίπεδο απορρόφηση για τη Ρουμανία νομίζω ότι είναι μηδέν όσον αφορά το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν νομίζω ότι έχουν αποσταλεί ε, κάποιοι λογαριασμοί στην, ε, στις Βρυξέλλες για να πληρωθούν για αυτή την περίοδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω μπει και εγώ στο κατάλογο των ομιλητών ε, για τη Ρουμανία. Να σας πω καταρχάς πως χαιρόμαστε για κάθε πρόοδο που επιτελείται η Επιτροπή μας έχει προσπαθήσει να συνοδεύσει τις προσπάθειες τόσο της Βουλγαρίας όσο και της Ρουμανίας στο διάστημα αυτών των ετών έτσι ώστε να γίνει καλύτερη χρήση των κονδυλίων. Ε, τώρα θα ήθελα να τοποθετηθεί ο κύριος Γενικός Διευθυντής και να μας πει γιατί ε, τι ακριβώς συμβαίνει με τα δικαιώματα των ε, κρατουμένων και τι ακριβώ γίνεται με αυτήν την κριτική που έχει ασκηθεί για το συνταγματικό δικαστήριο. Γιατί χρειάζονται 33 ε, τροπολογίες οι οποίες ε, θα ευνοήσουν περίεργο ποιου. Αυτό το συστημικό πρόβλημα είναι τεράστια δυναμία των ε, ταμείων. Σίγουρα όλοι θέλουμε να βελτιωθεί η κατάσταση έτσι ώστε η Ρουμανία να μπορέσει να ε, απορροφήσει και να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια, όμως πρέπει να ισχύει το ίδιο δίκαιο για τη Ρουμανία που ισχύει και στα υπόλοιπα κρατημέλη. Αυτή η συστημική πολιτική διαφθορά είναι σοβαρό πρόβλημα σε ορισμένα κρατημέλη. Γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν και λεφτές αυτές οι προσπάθειες που έγιναν και πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο, να δημιουργήσουμε τις σωστές προϋποθέσεις για να διορθωθεί ε, αυτό το πρόβλημα. Ο κύριος Ντόλτς έχει ζητήσει το λόγο και του τον δίνω αμέσως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γενικέ Διευθυντά, ήθελα να κάνω μια σύνοψη και να σας θέσω κάποιες ερωτήσεις. Καταρχάς, συμφωνείτε με αυτά που ακούσαμε για το μετρό της Βουδαπέστης από τον κύριο Γενικό Διευθυντή. Ε, αυτό είναι ένα έργο το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί κατά μεγάλο μέρος από κοινοτικούς πόρους. Και βλέπουμε λοιπόν στην έκθεση της Όλαφ ε, τι έχει γίνει. Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας μας έχει πει πως κάθε ευρώ, κάθε λεπτό που δαπανήθηκε πρέπει να ελεγχθεί και έχει ελεγχθεί και εμείς χρησιμοποιούμε την αρχή της μηδενικής ανοχής σε οποιοδήποτε φαινόμενο διαφθοράς. Όπως είπε και ο κύριος Γενικός Διευθυντής, τις τελευταίες εβδομάδες ε, είδαμε και έμπρακτα αυτό που λέμε. Οι έρευνες ε, δίρκησαν αρκετό καιρό. Η κυβέρνηση μάλιστα είχε αναλάβει και εκείνη ένα κομμάτι των ερευνών και μάλιστα όταν ε, βρέθηκαν οι πέτοι επιβλήθηκαν ποινές. Υπήρξαν αντιδράσεις βέβαια για αυτή την ε, πράξη της ε, κυβέρνησης. Το θέμα πήγε στα δικαστήρια. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Γενικές Διευθύνσεις και η Όλαφ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ε, συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει όμως κάποια σύγκρουση συμφερόντων ενδεχομένως και πρέπει να γίνει μια διερεύνηση της κατάστασης. διότι δεν γίνεται να γίνονται έκνομες ενέργειες χωρίς καμία ε, τιμωρία, χωρίς καμία ποινή. Και η κοινή γνώμη στην Ουγγαρία το συζητά αυτό και σίγουρα η κοινή γνώμη επηρεάζεται από τους πολιτικούς και από την, τις κομματικές γραμμές. Το 2010, ας πούμε, είχαμε μία κυβέρνηση συνασπισμού σοσιαλιστών και φιλελεύθερων, μετά έγινε μία τρικομματική κυβέρνηση και οι έρευνες της Όλαφ παρατήρησαν προβλήματα σε 30 διαφορετικές συμβάσεις. 30 συμβάσεις οι οποίες είχαν υπογραφεί αυτά τα χρόνια. 29 μάλλον, όχι όλες, 29 από αυτές τις 30 συμβάσεις είχαν υπογραφεί ε, όσο οι σοσιαλιστές βρίσκονταν στην κυβέρνηση της Ουγγαρίας. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή ένας διάλογος ε, που λαμβάνει η χώρα στην Ουγγαρία και η κοινή γνώμη σίγουρα έχει διαμορφώσει μία άποψη, γίνονται δηλώσεις και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω τον κύριο Γενικό Διευθυντή και την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Πολιοδομίας τι θα γίνει με την έκθεση, με τη δημοσίευση της. Δεν έχει γίνει μετάφραση στα ουγγρικά μέχρι τώρα. και έχουμε παρατηρήσει ότι κάθε φορά που η κυβέρνηση της ε, Ουγγαρίας ζητά λεπτομέρειες εξηγήσεις, λαμβάνουμε τελείως διαφορετικές πληροφορίες, τελείως διαφορετικές απαντήσεις. Ε, κάθε φορά που ζητάμε από την, γενική, από την αμμόδια γενική διεύθυνση κάτι μας απαντάει όλα. Είναι περιδεμένα τα πράγματα. Ε, ακούμε για, για θέματα ασφαλείας, για διάφορα τέτοια προβλήματα εξαιτίας των οποίων δεν μπορεί να δημοσιευθεί η έκθεση της Όλαφ. Όμως ε, όταν κάθε φορά που ένας ε, ευρωβουλευτής ή ένας βουλευτής ε, της Ουγγαρίας στέλνει μια επίσημη επιστολή στην Όλαφ ακούγονται διαμαρτυρίες. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντας την άποψη ότι αυτή η έκθεση πρέπει άμεσα να δημοσιευθεί στην ολότητά της για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Και να δούμε ακριβώς τι γίνεται στη συνεργασία των ε, Ουγγρικών Αρχών και της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για παράδειγμα. Θα ήθελα όμως να ακούσω και την άποψη του κύριου Γενικού Διευθυντή γι' αυτό. Τέλος, θεωρώ αρκετά σημαντικό η δική μας Επιτροπή να είναι πάρα πολύ προσεκτική με τις εκφράσεις που χρησιμοποιεί. Στην Ουγγαρία δεν υπάρχει συστημικό πρόβλημα, τουλάχιστον εγώ δεν έχω αντιληφθεί κάτι τέτοιο. Ιδιαίτερα μάλιστα από το 2014 και μετά, από το 2010 μάλιστα, Έχουμε αρχίσει να βλέπουμε αποτελέσματα στις προσπάθειες, όμως ε, σε ό,τι αφορά το, την γραμμή 4 του μετρό, η Όλαφ ε, διαπίστωσε κάποιες παρατυπίες και θέλουμε να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Γενικό Διευθυντή για αυτά που μας είπε. Ζούμε σε έναν πολιτικό κόσμο. Έρχονται και απέρχονται οι κυβερνήσεις και αλλάζουν συνεχώς. Το σημαντικό είναι όταν υπάρχει πρόβλημα που εντοπίζεται η τότε κυβέρνηση θα πρέπει να δείξει ότι κινείται για να διορθώσει την κατάσταση. Θα ήταν καλό να έχουμε μια απάντηση από την Ουγγρική κυβέρνηση και πληροφορίες όταν τελικά κινηθεί η κυβέρνηση. Να δούμε πώς καλύπτονται αυτά που θέσατε μετά την έκθεση Σόλαφ για τη Ρουμανία. Ήμουν στην Επιτροπή Ελέγχου, α, συγγνώμη, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης στη Ρέζη και εκεί είπατε ότι το ποσοστό απορρόφησης στη Ρουμανία είναι μηδέν. Και είπατε ότι ένα από τα προβλήματα είναι η μεγάλη δυσκολία εκπλήρωσης της ερεσιμότητας, της εκ των προτέρων ερεσιμότητας και στη Ρουμανία και στις χώρες. Είπατε ότι κάποια τεχνική αρρωγή έχει χορηγηθεί και μάλλον θα ξεκινήσει πολύ γρήγορα. Τα πρώτερα προβλήματα που θέσατε για τον έλεγχο προπολογισμού, ότι δεν μπορείτε ακόμα να καθορίσετε ένα σύστημα ελέγχου, συνδέονται αυτά. Από τη στιγμή που η τεχνική αρρωγή θα παρασχεθεί, θα δούμε κάποια επίπεδα απορρόφησης και θα δαπανώνται οι πόροι. Θα βελτιωθεί επίσης και το σύστημα ελέγχου. Συνάδελφε Τσέλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είχα μία πρόταση για την ε, νομοθεσία και για τους νομοθέτες της ε, κυβέρνησης. Σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις διαφθοράς βλέπουμε, θα ήθελα να προτείνω ένα πρόστιμο ύψους 50, μέχρι 50.000 ευρώ. Αυτό για άτομα τα οποία ήδη έχουν καταδικαστεί για περιπτώσεις διαφθοράς. Θα έχουν λοιπόν την δυνατότητα, δεν θα πρέπει να έχουν μάλλον, τη δυνατότητα να διεκδικούν μετά πολιτικά αξιώματα όσοι έχουν καταδικαστεί για διαφθορά. Η επικεφαλής της ε, υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς, κυρία Κόβασιτ, είπε πως Εάν είχε τεθεί σε εφαρμογή αυτός ο νόμος θα μπορούσαν να είχαν κερδίσει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ με κατασχέσεις από τέτοιες περιπτώσεις ε, καταδίκης για διαφθορά. Εσείς τώρα θα ήθελα να ρωτήσω ε, τι προβλέπετε να γίνει από εδώ και στο εξής. Έχουμε ένα μέλος του Κοινοβουλίου και μάλιστα έναν από τους πλουσιότερους ε, ανθρώπους της Ρουμανίας που έχει αρχίσει μία εκστρατεία πολέμησης της διαφθοράς. Ε, και το έργο αυτό έχει απολαύσει την ε, θετική γνώμη του κοινού. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες περιφερειοποίησης αν θέλετε, καλύτερης χρήσης των κονδυλίων, ανεξάρτητα από το που ανήκει πολιτικά όποιος ε, βρίσκεται σε ηγετική θέση την εκάστοτε στιγμή. Εάν λοιπόν γίνει αυτή η περιφερειοποίηση στη χώρα, τότε ίσως θα πληρούταν και μία από αυτές τις προϋποθέσεις ε, βελτίωσης της διοίκησης. Θα μπορούσατε λοιπόν να εξετάσετε μια τέτοια πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γενική Διευθυντά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ξεκινούσα με το συγκεκριμένο ερώτημα του κυρίου Ιβεν για τις προπτικές που υπάρχουν, ούτως ώστε η Ρουμανία να ξεκινήσει την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτής της περίοδου. Άρα με αυτή την απάντηση θα δώσω και κάποια στοιχεία απαντήσεως σε αυτά τα ερωτήματα του κ. Βόβεν. Έχουμε δύο ξεχωριστά ζητήματα. Το πρώτο, η διαδικασία καθορισμού συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης. Πάνω σε αυτό η Ρουμανία θα έλεγα ότι αντιμετωπίζει περισσότερο τεχνικά προβλήματα και όχι διαρθρωτικά. Ούτε προβλήματα διοικητικού δυναμικού. Τα τεχνικά προβλήματα συνδέονται με τα νέα συστήματα πληροφορικής που χρειάζεται να δημιουργηθεί. Και αυτό το πρόγραμμα για την πληροφορική έχει καθυστερήσει και κατά πολύ. Θα έλεγα ότι εν γέννη, αν δεν υπήρχε αυτό το στοιχείο, οι προοπτικές θα ήταν σχετικά καλές. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία για τον καθορισμό των συστημάτων. Συνοδεύουμε όσο καλύτερα μπορούμε την Ρουμανία στις προσπάθειές της. Και τη νέα κυβέρνηση τώρα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν τα αναπομένοντα προβλήματα. Ο καθορισμός ε, είναι προαπαιτούμενο για την καταβολή πληρωμών. Μπορούν να γίνουν πράγματα όμως για να προχωρήσουμε προς την υλοποίηση τα οποία δεν απαιτούν αναμονή για ολοκλήρωση αυτού του βήματος. Δεν σημαίνει ότι θα ήταν αδύνατον η Ρουμανία να προχωρήσει με την επιλογή προγραμμάτων. και βλέπουμε αυτό σταδιακά να πραγματοποιείται. Ε, δεύτερον, αυτό που προανέφερα. Οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες. Οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες είναι όροι που ορίζονται σε διάφορους τομείς. Οι προποθέσει αυτέ που καθορίζονται, αν δεν εκπληρώνονται μέχρι κάποια χρονική στιγμή, μπορεί να οδηγήσουν σε αναστολή πληρωμών. Στην περίπτωση τη Ρουμανία, το πρώτο εμπόδιο είναι ο καθορισμό, να μπορεί να υποβάλει πληρωμέ, αιτήσει πληρωμών η Ρουμανία. Μετά όμω έρχεται ένα δεύτερο στάδιο, δεύτερο έλεγχο, για την εκπλήρωση των εκ των προτέρων ρεσιμοτήτων. Και όσον αφορά αυτό, Χρειαζόμαστε κάποια πρόοδο σε έναν τομέα και έχει πληρωθεί μεγάλη πρόοδος μέχρι τώρα, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα και είναι ο τομέας ε, των κρατικών προμηθειών. Εκεί θα παραμείνουμε πάρα πολύ απαιτητικοί. Όμως είμαστε στο σωστό δρόμο και περιμένουμε τελικά ότι αυτή εκ των προτέρων αιρεσιμότητα θα μπορεί να καλυφθεί αν όλα πάνε καλά μέχρι, το τέλ, μέχρι τα μέσα μάλλον ενεστώτος έτους. Τώρα για τα δύο σχέδια διαταγμάτων. Να πω ξανά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί εκ του ε, τις εξελίξεις και μαζί με αυτά που σας προανέφερα, δηλαδή συγκεκριμένες αναφορές για τις πρόσφατες εκθέσεις για την ε, Ρουμανία βάσει του μηχανισμού CDM και με την ανοιχτή αιμονή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα πρέπει να αποδειχθεί ότι η πρόοδος είναι αμετάκλητη. Ε, αυτά είναι σαφή μηνύματα που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα παρακολουθούμε πάρα πάρα πολύ προσεκτικά τις εξελίξεις. Και υποθέτω ότι σύντομα, πολύ σύντομα θα υπάρξει δυνατότητα ο ίδιος ο κύριος Τίμερμανς να προβεί σε ανταλλαγή απόψεων με τους κοινοβουλευτικούς φορείς για το συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Ντόιτς, νομίζω σωστά περιγράψατε συμπληρώνοντας με την κατάσταση. Πράγματι θεωρούμε τώρα ότι έχουν ξεκινήσει διάφορες νομικές διαδικασίες από τις Ουγγρικές αρχές. Ακριβώς γι' αυτό εμείς δεν μπορούμε να αποφασίσουμε και δεν αφορά τη διεύθυνσή μου, τη Γενική Διεύθυνση Ρίτζο εξάλλου, διότι είναι έκθεση της Όλαφ, γι' αυτό έλεγα δεν μπορούμε να αποφασίσουμε ε, τη δημοσίευση της εκθέσεως. Και γι' αυτό η απόφαση για αυτή τη δημοσίευση είναι κάτι που αφορά τις Ουγγρικές Αρχές τώρα, διότι οι Ουγγρικές Αρχές είναι εκείνες που γνωρίζουν το περιεχόμενο των ε, εθνικών αυτονομικών διαδικασιών και γνωρίζουν ποια θα μπορούσε να είναι η μορφή της εκθέσεως όταν θα εκδοθεί με το σεβασμό της προστασίας ιδιωτικών στοιχείων βεβαίω. Αυτό το θέμα μερικής δημοσιοποίησης της εκθέσεως είναι κάτι που αφορά την α, ε, ε, ουγγρική κυβέρνηση, τις ουγγρικές αρχές. Τέλος, κύριε Βόν, ελπίζω να διευκρίνησα κάπως ποια είναι η φύση του μηχανισμού καθορισμού και μετά ε, κάπως και τη φύση των εκ των προτέρων ρεσιμοτήτων. Και τέλος, κύριε Τσέλερ, να απαντήσω και σε εσά. Η Κομισιόν δεν έχει βέβαια αρμοδιότητα να αποφασίσει ε, για την ε, δαφική οργάνωση των κρατών μελών. Εντάξει, βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων με τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή των διαφορών επιχειρησιακών προγραμμάτων, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε πως η προσέγγιση θα είναι η καλύτερη δυνατή, ως προς τα αποτελέσματα φυσικά. Για παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα το περιβάλλον. Αυτό που φαίνεται να είναι εκ των όνου ουκάνευ. Για μας είναι μια καλή συνεργασία. Όπως βλέπετε, είπατε και εσείς σήμερα, στη Ρουμανία υπάρχουν ελάχιστα στάδια ανάμεσα στους δήμους, στις κοινότητες και στην κυβέρνηση. Σε επίπεδο όμως ε, τοπικό είναι πολύ σημαντικό οι δαπάνες ε, να είναι αποτελεσματικές, για παράδειγμα ε, διάφορα διάφορες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, λιμάτων και να γίνονται διάφορα κοινά έργα για να υπάρχει αυτή η κριτική, αυτή η κριτική μάζα. Αυτό δεν είναι κάτι που συναντούσαμε συχνά στο παρελθόν, όμως είναι μία εκ των προτέρων αρισιμότητα. που βασίζεται όχι στο επίπεδο συνεργασίας, αλλά στο υφιστάμενο διοικητικό σύστημα της Ρουμανίας. όπου βλέπουμε ότι σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης υπάρχουν άλλοι παράγοντες. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις σημαντικότατες πληροφορίες. Είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε ε, και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κρατη ότι έχουμε μία εποπτεία της κατάστασης. Γιατί διάβαζα μάλιστα πρόσφατα ότι σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Ουγγαρία, ε, μετά από την ε, δημοσίευση της έκθεσης υπήρξαν διάφορα προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν σε εμά είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι γίνεται Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας κρατήσετε ενήμερους για το τι γίνεται στην, Ουμαρία, στη, στην Ρουμανία. Στη Ρουμανία θα παρακολουθήσουμε και εμείς βέβαια πολύ στενά την κατάσταση. Αλλά θα ήθελα να κάνω μια παράκληση η Κομισιό να μην καταβάλει αυτά τα κονδύλια. Κάτι που με λυπεί πάρα πολύ διότι τα έχει ανάγκη. Αλλά μέχρι να λυθούν αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να γίνει αναστολή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και που μας ενημερώσατε για την κατάσταση. Εμείς ως Επιτροπή Ελέγχου του προπολογισμού, σίγουρα θα είμαστε ενήμεροι και θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Εδώ διακόπτω τη συνεδρίαση μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Ευχαριστώ.